Buenas tardes. Reanudamos la, la sesión. Καλό σας απόγευμα. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση εκ νέου. Με πολύ μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Γεωργία Τροφιμών και Ναυτιλία τη ε, Ιρλανδία, στον οίκο του και στην Επιτροπή του. Είναι παλιό ε, γνωστό σα. Ήταν μέλο αυτού του κοινοβουλίου και αναπληρωτικό μέλο τη Επιτροπή Αλία. Και Νομίζω ότι πέρα από την ε, κανονική φιλοξενία που έχουμε με τους εκπεριτροπείς ε, υπουργούς, ε, έχουμε και προσωπική φιλία με έναν άνθρωπο που είναι πιο κοντά σε αυτή την επιτροπή. Έχουμε μία πιο κοντινή σχέση σε αυτή την περίπτωση. Και θα έλεγα ότι ο κύριο Υπουργό γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει διαφορετικά καθήκοντα. Επίσης, ε, θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την παρουσία του, αλλά και για τη δυνατότητα που είχαμε να, γευματίσουμε, να προγευματίσουμε μαζί την περασμένη εβδομάδα μαζί με τους συντονιστές. Άτυπο ήταν αυτό το πρωινό, αλλά μπορέσαμε να αναλύσουμε ορισμένα από τα θεμελιώδη προβλήματα που συζητούμε σε αυτή την επιτροπή. Πρόκειται για μια μικρή επιτροπή, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Και τότε το είχαμε ζητήσει, αλλά τώρα το επαναλαμβάνω και επίσημα. Έχουμε μια πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ένα από τα κυριότερα θέματα είναι με τα τη κοινή ελευθερική πολιτική που έχει προχωρήσει. Ήδη ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο το βασικό κανονισμό. Και τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Καντέικ επί τη ουσία και έχει προβλεφθεί ψηφοφορία για το Μάρτιο. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση για την οποία όλοι έχουμε πολύ μεγάλες ελπίδες, είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει για κάποια στοιχεία, όπως είναι τα σχέδια διαχείριση. σημαντικό τμήμα αυτή τη μεταρρύθμισης και είναι το μεγάλο εμπόδιο που μας διαχωρίζει από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει μια θέση αντίθετη με αυτή την ε, νομική υπηρεσία, με όσα λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που μας εκχωρεί η συνθήκη. Και εγώ θέλω να δηλώσω εδώ δημόσια ότι αυτό είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές να αναλάβει ο Υπουργός για το εξάμενο αυτό, αν θα καταστεί κανός, να άρει αυτά τα εμπόδια για να απεμπλοκαριστεί η κατάσταση σε σχέση με τα σχέδια διαχείρισης. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε από κοινού προς την διακατεύθυνση. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση, αλλά επίση ε, γνωρίζουμε τι ικανότητε του Υπουργού και τι γνώσει που έχει. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα και το Συμβούλιο, βέβαια, για να προσπαθήσει να μα βοηθήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν φυσικά και άλλα θέματα που θέτουμε, όπω είναι η εξωτερική διάσταση τη κοινή ελευτική πολιτική, οι συμφωνίε, είναι πολύπλοκε αυτή τη στιγμή, λίγε συμφωνίε και κάποιε υποδιαπραγμάτευση δύσκολη. Έχω κατά νου αυτή με το Μαρόκο και όπως ε, για την κατάσταση με τη Μαυριτανία. Και νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές και σίγουρα δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος μπροστά σας για τον τομέα της Ελίας στο εξάμεινο αυτό. Εμείς βέβαια όπως σας είπα περιμένουμε πολλά. Δεν θα μακρηγορήσω, επομένως θα αφήσω το λόγο στον κύριο Υπουργό και πάλι να τον ευχαριστήσω και να επαναλάβω την επιθυμία μας ε, να πετύχει γιατί αν πετύχετε θα πετύχουμε κι εμείς. Έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. And, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να είμαι και τυχερός. Καλύτερα να είναι τυχερός ο στρατηγός παρακαλώ. καλός. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα πρόσφατα ήταν, που καθόμουν ε, στη θέση του βουλευτού, του μέλους της Επιτροπής, αυτή την αίθουσα. Είναι προνόμιο για μένα να μην είμαι από την άλλη πλευρά του τραπεζιού κατά την ελλανδική Προεδρία. Ελπίζω όμως, λόγω της εμπειρίας μου εδώ, επί τρία χρόνια, και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και σαν ένα πληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αλίας ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε προσπαθώντας να σημειώσουμε σημαντική αν όχι πλήρη ε, μεταρρύθμιση της κοινής αδιευτικής ε, πολιτικής. Αυτή είναι η φιλοδοξία της Προεδρίας μας σχετικά με το θέμα και ελπίζω να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και ξεκάθαρης ομή συζήτηση που είναι απαραίτητη ούτως ώστε από κοινού να προωθήσουμε το πρόγραμμα αυτό και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Βέβαια, δουλειά μου είναι σαν Προεδρεύον του Συμβουλίου να εκπροσωπώ τη θέση του Συμβουλίου. Επίσης, όμως, θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας για την εξέβρεση λύσεων, απαντήσεων και συμβιβασμών. για τις προτεραιότητες που ξέρω ότι έχετε σαν Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή. Χαίρομαι, όπως προανέφερα, που είμαι εδώ και συναντώ με στην ε, Επιτροπή αυτή σαν προεδρεύων του Συμβουλίου ε, Αλίας. Είναι η 7η Προεδρία της Ιρλανδίας και είναι η 40η επέτειος της προσχωρήσεως της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ε, είναι η πρώτη φορά που λειτουργούμε βάσει τη συνθήκη τη Αβώνα που έχει εισαγάγει σημαντικέ νομοθετικέ αλλαγέ όσον αφορά ε, τι εργασίε, τη εξαγωγή των εργασιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, κυρίω όσον αφορά την κοινή πολιτική. Στα πλαίσια λοιπόν τη Προεδρία μα, Είμαστε οι πρώτοι από, ένα τρίο. Θα ακολουθήσει η Λιθανία και η Ελλάδα μετά. Το γενικό θέμα της Προεδρίας της Ιρλανδίας είναι ένα πρόγραμμα πολιτικών που εστιάζεται με τις λέξεις σταθερότητα στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Είναι ένα πρόγραμμα εργασίας με κέντρο τους ε, ανθρώπους και την ανάκαμψη και σε κάθε τομέα πολιτικής στα εννέα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ενώσης, των οποίων προεδρεύουμε σαν Προεδρία, θέλουμε να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις και να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος και δεν αποτελεί εξαίρεση το μέσα αλίας. Ε, είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε να επενδύσουμε σε ανάπτυξη που είναι φιλική και θέλουμε να